και μπορούμε να περάσουμε στην ώρα των ερωτήσεων. Η πρώτη ερώτηση είναι η παριθμό 15. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στο χρόνο γιατί 8.30 πρέπει να ολοκληρώσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι της, της κυρίας Γκουτιέρες Κορτίνες. Την αναπληρώνει εδώ ο κύριος Γκαρίγκα Πολέντο. Θα ακούσουμε πρώτα την απάντηση της Επιτρόπου. Κυρία Γεγενκού είναι όποτε Είστε εύκαιροι, μπορείτε να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ. Το πρώτο τμήμα της ερώτησης κυρίας Γκουτιέρες Κορτίνες αφορά το κατά πόσο τα κριτήρια επιλογή για το ανώτατο διοικητικό προσωπικό των καιρών τεχνολογικών πρωτοβουλειών εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του από την επιρροή των μεγάλων επιχειρήσεων. Η απάντηση είναι καταφατική. Η... Τα κριτήρια επιλογή ε, των στελεχών ακολουθεί τι κατευθυντήριε γραμμέ που ισχύουν για όλα τα κοινοτικά όργανα και εξασφαλίζουν ότι η, επιλογή, ε, η διαδικασία επιλογής για τις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες είναι αντίστοιχη με τις επιλογές σε άλλες ρυθμιστικές ή κανονιστικές αρχές. Ακόμη και για τις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες, τα κριτήρια επιλογής είναι αξιοκρατικά και εξασφαλίζεται η συμμεταχείριση όλων των υποψηφίων. Από την άποψη αυτή, όπως προβλέπετε και στις κατευθυντήριες γραμμές, ψηλόβαθμη υπάλληλη της Επιτροπής είναι επιλογή και στην φάση της προεπιλογής, αλλά και κατά την τους διορισμούς. Αυτά είναι μόνο τα δύο στάδια που και ο κλάδος είχε ένα ρόλο. Πέραν του έμεσου ρόλου κατά την ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη στιγμή της, ε, του διορισμού. Μετά από το κατάλογο που έχει προεπιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, το κόστος ε, διαχείρισης των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών καλύπτονται σε επίπεδο 67% από τον κλάδο. Επίσης, οι δύο κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες για τις νανοτεχνολογίες και τα σωματωμένα συστήματα υπολογισμών ακολουθούν αυτόν τον κανόνα. Εξασφαλίστηκε η απαραίτητη συμμετοχή και διασφαλίστηκε και ο χαρακτήρας των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών ως συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και φορέων. Τώρα, κατά πόσο ε, λήφθηκε υπόψη και το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα κριτήρια επιλογή ε, του προσωπικού για την καθημερινή λειτουργία των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών θα πρέπει να πληρεί τι κατευθυντήριε γραμμέ για το διορισμό που ε, εφαρμόζουν αξιοκρατικά κριτήρια. Η προαγωγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντικό πολιτικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν μπορεί να μεταφραστεί σε κριτήρια επιλογή για το διορισμό προσωπικού που καλύπτονται από του ε, κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα και για το προσωπικό των κοινών τεχνολογικών πρωτοβουλειών. Ισχύουν εδώ και Επαγγελματικέ αρχές, οπότε δεν ε, εκπροσωπούνται ιδιαίτερα συμφέροντα ούτε μικρομεσαίων επιχειρήσεων ούτε μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Προβλέπονται επίση κάποιε πειθαρχικέ διαδικασίε για παραβιάσει αυτών των διοντολογικών κριτήριων. Ο κανονισμό, βέβαια, που θεσπίζει τι κοινέ τεχνολογικέ πρωτοβουλίε, ε, προβλέπει κάποιε διατάξει για την ε, ενθάρρυνση και προώθηση τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα διοικητικά συμβούλια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκαρίγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμμερίζονται τις ανησυχίες. Ε, κυρία Επίτροπε, όμως ε, η πράξη μας φάζει στην αντίθετη πορεία. Γνωρίζουμε ότι οι κοινές τεχνολογικές ε, πρωτοβουλίες έχουν ένα πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να γίνεται σεβαστό. Και δεν θα πρέπει τα άτομα να προέρχονται από επιχειρήσεις ή από άτομα τα οποία είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τα ειδικό, την κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για το υδρογόνο με προπολογισμό 470 εκατομμύρια ευρώ, κατάληξαν ε, σε ένα άτομο μεταξύ τριών τελικά. Πρόκειται για έναν ε, εμπειρογνώμονα που προέρχεται από μικρομεσαία επιχείρηση και όταν ε, τελικά έφτασε και να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαταστάθηκε από μέλος της Toyota Daimler, από μια στέλεχος μεγάλης επιχείρησης. Νομίζω ότι αυτό αντιβαίνει ε, σε αυτό που είπατε στην αρχή που θα πρέπει να είναι και η λογική η οποία θα διέπει αυτή τη διαδικασία. Ε, θα ήθελα λοιπόν να επαρρυπνείτε και να παρακολουθείτε κύριε Επίτροπε, τη διαδικασία επιλογής. Πρόεδρος. Ξέρετε ότι μισό είναι το λεπτό μόνο για τη δευτερολογία, αλλά τέλος πάντων η Επίτροπος θα ήθελα να απαντήσει. Βεβαίως. Θα επαγρυπνώ, όπως μου ζητήσατε, για αυτό το θέμα και νομίζω ότι πρέπει να σημειωθεί ότι τα έξοδα διαχείρισης καλύπτονται εν από τον κλάδο και σύμφωνα με τη συμβολή αυτή και με το πνεύμα των συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα γίνονται, ε, προβλέπονται κάποια πράγματα για το διορισμό των μελών των νοικητικών Συμβουλίων. Σίγουρα ε, το συμβούλιο, το, υπάλληλοι ε, της Επιτροπής είναι πάντα πλειοψηφία στη δικασία επιλογής. Ο κλάδος συμμετείχε με δύο τρόπους και ίσως ε, θα ήταν ε, καλό να σας πω πώς λειτουργεί. Ένας στους τρεις από την Επιτροπή Προεπιλογής έχει δικαιώματα ψήφου και ο άλλος είναι διευθυντής, γενικός διευθυντής ή αναπληρωτή γενικό διευθυντή, προεδρεύει αυτός και υπάρχει επίση ε, και ένας ε, διευθυντή. Υπάρχει παρατηρητή επίση συμβουλευτική επιτροπή για του διορισμούς που δεν έχει όμω δικαίωμα ψήφου και μετά από τα έξι ε, μέλη επιλογή της συμβουλευτική επιτροπή είναι μέλη τη Επιτροπή Τρει στου έξι σε ό,τι αφορά τη το συγκεκριμένη κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία που είπατε προέρχονται από μικρομεσαία επιχείρηση. Και αυτό ότι πρέπει να προέρχεται δηλαδή από την μικρομεσαία επιχείρηση το λέει και το καταστατικό της κοινή αυτής της τεχνολογικής πρωτοβουλίας. Βεβαίω πάντως και θα επαγρυπνώ, όπως μου ζητήσατε, κύριε Βουλευτά, για τις μελλοντικές τέτοιες διαδικασίες. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στο ερώτημα 16 της κυρίας Σένισιν. Αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να καθίσει ο Επίτροπος για να απαντήσει. ready, Κύριε Σέμιτα, όταν είστε έτοιμος έχετε το λόγο. Honorable member, η προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών δεν θα επηρεάσει ε, τον τρόπο ε, δράση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, και των πρόσφυγων κατά οποιασδήποτε χώρα. Η προσχώρηση θα δημιουργήσει κάποιες υποχρεώσεις με βάση τη συνθήκη και θα εφαρμοστεί οποιοδήποτε συμπληρωματικό πρωτόκολλο που θα επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά μέτρα και δράσεις που υιοθετούν οργανισμοί, αρχές ή θεσμικά όργανα της Ένωσης. Αλλά δεν αφορά μέτρα που έχουν θεσπιστεί και εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Ούτε προβλέπεται η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομολογίας του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί δεν υπάρχει νομική βάση για τη θέσπιση ενό τέτοιου μηχανισμού. Το πρωτόκολλο υπαριθμών 8 τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα απαιτεί ε, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, να μην επηρεάζει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα την κατάσταση των κρατών μελών σε σχέση με την σύμβαση. Αυτό αφορά όχι μόνο το πεδίο εφαρμογή των ουσιαστικών υποχρεώσεων των κρατών μελών, αλλά αφορά και τον τρόπο με τον οποίο μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά μια ε, ευρωπαϊκή χώρα εκτελείται. Σα ευχαριστώ για τη συμπληρωματική ερώτηση. Η κυρία Σένισιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Επίτροπο για την απάντηση. Δυστυχώς δεν με ικανοποιεί η απάντηση αυτή, γιατί ο έλεγχος της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι απαραίτητος. Γιατί φαίνεται ότι ε, κάποιες χώρες δεν θέλουν και οθελώς να εφαρμόσουν αυτή την ομολογία, αυτές τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Σε ό,τι αφορά ε, την απόφαση κατά της Ιταλίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε την ε, απόφαση για την ε, παρουσία του σταυρωμένου της τάξης ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης υπήρξε κάποιο θέμα με το μάθημα των θρησκευτικών. Οι νομικές αυτές διατάξεις που, της Πολωνίας που κατηγορήθηκαν ως παράνομες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυρία Σένισιν, ε, ακούσαμε την συμπληρωματική σας ερώτηση. Νομίζω ότι ο Επίτροπος κατάλαβε περί την πρόκειται και μπορεί να απαντήσει. Ε, ε, Θα προσπαθήσω να απαντήσω Όταν τα κράτη-μέλη δρούν στα πλαίσια του ενωσιακού νόμου θα πρέπει να τηρούν τον χάρτη και τις γενικές αρχές του ε, ε, ενωσιακού δικαίου και οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της υποχρέωσης οδηγεί σε διαδικασία επιπαραβάση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει άρθρου 258 της Συνθήκης Λειτουργίας Ένωσης τι είναι η μόνη διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την συμμόρφωση κράτους μέλους με θεμελιώδη δικαιώματα. Αντίθετα, όταν κινούνται εκτός του ενωσιακού δικαίου τα κράτη-μέλη, αλλά δεν υπάρχει γενική αρμοδιότητα βάσει συνθήκων ε, στον τομέα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ένωση παρακολουθεί το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα κράτη-μέλη και αν συμμορφούνται ε, προς τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δύο συμπληρωματικές μαζί. Πρώτα ε, η κυρία Γκέρντιν και μετά η Λέδη Λάντφορντ. Μισό... Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα θα συμμετέχει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση. Από τα σημαντικότερα θέματα θα είναι οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του ΔΕΚ. Πώς ε, θα εξασφαλίσετε ε, τη διασφάλιση των αρμοδιοτήτων του ΔΕΚ σε ό,τι αφορά την ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου. Ευχαριστώ. Η Βαρόνι Λάτφορτ. Από τεχνική και νομική άποψη αντιλαμβάνομαι την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από πολιτική άποψη όμως και από άποψη προσήλωση στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τελείως παράλογη και παρανοϊκή η απάντηση και ε, υπονομεύουν το άρθρο 6 και 7 της συνθήκης που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα τηρήσουν το μηχανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και υπάρχει μηχανισμό ε, στο άρθρο 7 για να αποφευθεί η καταστρατήγηση των διατάξεων για τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Πώ πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει συμβατότητα με το άρθρο 7. Χρειαζόμαστε μηχανισμό εποπτεία και ελέγχου. Και φάνηκε η αδυναμία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ασκήσει προσφυγή κατά κρατών μελών σε περίπτωση καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, uh, uh, Ακούστε. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τις διαπραγματεύσεις ότι ο στερικός έλεγχος ε, του ΔΕΚ ε, με βάση το πρωτογενές δίκαιο θα εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου η συμμόρφωση ενός θεσμικού οργάνου ή φορέα ε, με τη σύμβαση τίθεται υπό αμφισβήτηση και επομένως θα πρέπει να επιλαμβάνεται το 10. Σε ό,τι αφορά όμως τη συμβατότητα συγκεκριμένης πράξης ε, με ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν έχει αρμοδιότητα το ΔΕΚ. Θα πρέπει όμως το ΔΕΚ να μπορεί να αξιολογεί τη συμβατότητα γιατί αυτό είναι σημαντικό όμως θα πρέπει να γίνεται υπόψη, να λαμβάνεται υπόψη και η αρχή της επικουρικότητας και δεν θα πρέπει να προκύπτουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, αλλά παρόλα αυτά σας ευχαριστούμε. Θα πρέπει να απαντηθούν οι ερωτήσεις μου. Οι δικές μου ερωτήσεις για το άρθρο 6 και 7, κύριε Επίτροπε, δεν το απαντήσατε σε σχέση με αυτά που είπατε και με τον μηχανισμό για την αντιμετώπιση διάφορων παραβάσεων. Ο Επίτροπος θα μπορούσα να σας ενημερώσω ότι συνεχίζεται το έργο στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε σχέση με κάποιες αποφάσεις ε, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή το έργο αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Μακάρι να μην καθυστερήσει πολύ, λέει ο πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε. Now στην επόμενη ερώτηση που είναι του κυρίου Παπα-Νικολάου και πάλι ο Επίτροπος Σέμετα θα απαντήσει. Ερώτηση υπαριθμό 17. Αξιότιμη κύριε Ευρωβουλευτά, επιβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πέρυσι στο Συμβούλιο μία πρόταση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών ε, και του πριγκιπάτου του Λίχτενστάιν για την καταπολέμηση της απάτης και οποιοδήποτε παράνομης δραστηριότητας και να εξασφαλίσει ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο ένα σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ανδόρα, το, το Μόνακο, το Σαν Μαρίνο και την Ελβετία το σχέδιο συμφωνίας και το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής εκκρεμούν αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο γιατί ορισμένα κράτη-μέλη έχουν πολιτικές επιφυλάξεις για τη διασύνδεση των δύο περιπτώσεων σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις αποταμιεύσεις. Θεωρώ ότι τα σχέδια αυτών των συμφωνιών και της ε, διαπραγματευτικής εντολής θα πρέπει να κρατηθούν εχμάλωτοι της ε, ε, οδηγίας και από τη στιγμή που χρειάζεται να προασπίσουμε τα κοινά χρηματοοικονομικά μας συμφέροντα και να πατάξουμε τη φοροαποφυγή, καλό θα ήταν να σημειώσουμε πρόοδο. Ορισμένες χώρες ε, ε, εποφελούνται από τους φορολογικούς παραδείσους ε, και τις offshore εταιρείε. Πάντως εγώ πιστεύω ότι οι προτινόμενε συμφωνίε θα συμβάλλουν στη βελτίωση της μεταβίβασης και ταλλαγή τέτοιου είδου πληροφοριών για φορολογικά θέματα και θα προωθήσουν την χρηστή διακυβέρνηση στα φορολογικά θέματα με βάση τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ανταλλαχής ε, πληροφοριών και του θεμητού φορολογικού ανταγωνισμού. Στόχος της πολιτικής αυτής δεν είναι μόνο να πατάξει τους φορολογικούς παραδείσους, αλλά να συνάψει συμφωνίες με όσο το δυνατό περισσότερες τρίτες χώρες με βάση τις κοινέ αρχές της συνεργασίας και της διαφάνειας. Το Συμβούλιο Εκοφήν αστερνίστηκε αυτές τις αρχές και αναγνώρισε την ανάγκη προαγωγής των αρχών αυτών σε όλο και πιο ευρεία γεωγραφική βάση. Και το σχέδιο συμφωνίας με το πρικυπάτο του λίχτεσταν και τη διαπραγματευτική εντολή για σύναψη συμφωνίες με άλλες χώρες αποτελούν ε, ε, πρωτοφανέ παράδειγμα τέτοια διεθνού συνεργασία και προβλέπουν ελάχιστου κανόνε για την ανταλλαγή πληροφοριών και αρρωγή μεταξύ των εταίρων και των, διαφόρων φορέων, ώστε να παταχθεί η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή με αποτελεσματικό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει και να προαγάγει την πολιτική διαφάνεια ανταλλαγή πληροφοριών και θεμητού φορολογικού ανταγωνισμού στη σχέση με τι τρίτε χώρε. Κάτι τέτοιο επιτυχάνεται μέσω πρωτοβουλειών όπως η διεύρυνση της διοικητικής συνεργασίας, δεοντολογικός κώδικας για τη φορολογία των επιχειρήσεων ή συνεργασία σε φορολογικά θέματα με αναπτυσσόμενες χώρες και η προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης σε φορολογικά ζητήματα που είναι σημαντικό στομέα των σχέσεών μας με τις τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης δραστηριοποιείται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και σε διεθνή, ε, διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο ΩΣΑ και το Παγκόσμιο Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών προ, προσπαθώντας να προωθήσει αυτή τη νέα διαδικασία. Σας ευχαριστώ κύριο Παπα-Νικολάου για συμπληρωματική ερώτηση. Μισό λεπτό. Κύριε Επίτροπε, προκύπτει από την πράξη αλλά και από όσα μας είπατε σήμερα ότι τα κράτη μέλη μόνο με τους δικούς τους ελεκτικούς μηχανισμούς δεν μπορούν αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν αυτό το σημαντικό πρόβλημα. και βεβαίως είναι δεδομένο ότι αυτή τη μορφή η φοροδιαφυγή επιφέρει σοβαρότατο πλήγμα στην ανάπτυξη και δημιουργεί ροές κεφαλαίων όχι με κριτήριο την απόδοσή τους αλλά πώς θα υπάρχει καλύτερη φοροδιαφυγή. υπάρχει και η άλλη προσέγγιση αυτή που υιοθετείται στην ιαπωνία στι ηνωμένε πολιτείε όπου η έλεγχοι στι καταθέσεις είναι πιο χαλαρή και ε, έτσι γίνονται λιγότερο ελκυστική η παράδειση η φορολογική αυτή παράδειση. βεβαίω σε κάθε περίπτωση αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κράτη μέλη που δεν έχουν αποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού γιατί θα επιφέρει απώλεια εσόδων. ρωτώ λοιπόν ποιε είναι οι προτεραιότητε τη επιτροπή ποια η στρατηγική τη ποιο είναι το δικό τη ε, μονοπάτι για αυτή την προσπάθεια και ποιες οι που θέλει να κρατήσει. Ε, συγγνώμη, νομίζω ότι γίνεται σαφής. Θα απαντήσει ο Επίτροπος τώρα. Καταρχήν να πω ότι όταν διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες, αυτές που ανέφερα, διαπραγματευόμαστε εξ ονόματος των 27. Είναι πολυμερής η προσέγγιση. Όταν διαπραγματευόμαστε θέματα που αφορούν τη φοροδιαφυγή. Είναι ενδιαφέρον το θέμα αυτό και όντως εξετάζουμε διάφορους τρόπους αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής με τις μορφές που παίρνει και πολύ σωστά είπατε ότι οι φοροδιαφεύγοντες προσαρμόζονται στις αλλαγές των ελέγχων των δικών μας. Γι' αυτό έχουμε αυτή την ομάδα κώδικα δεοντολογίας όπου προσπαθούμε να ε, την εφαρμόσω, να τον εφαρμόσουμε όχι σε επίπεδο κρατών μελών μόνο, αλλά θέλουμε να ενθαρρύνουμε και τρίτες χώρες να σπαστούν αυτόν τον κώδικα ή τουλάχιστον να σπαστούν κάποιες αρχές του κώδικα αυτού. Έτσι θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε πρόοδο στον τομέα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ. Δύο συμπληρωματικές μαζί. Ζέμκε και Κέλλη. Ο κύριος Ζέμκε, 30 δευτερόλεπτα. Έχω και εγώ μια ερώτηση κύριε Επίτροπε. Από ό,τι μας είπατε, έχουμε ένα πολύ καλό σχέδιο, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί το μπλοκάρει μια ομάδα κρατών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορείτε να κατονομάσετε συγκεκριμένες χώρες. Πόσες όμως είναι αυτές οι χώρες που εναντιώνονται στο σχέδιο αυτό και τι επιχειρήματα επικαλούνται για να τεκμηριώσουν την αντίθεσή τους. Γιατί κάποιου λόγου θα πρέπει να έχουν αυτέ οι χώρε που είναι διστακτικέ απέναντι στο σχέδιο. Ποια είναι τα επιχειρήματά του, ο κύριο Κέλλη. Άκουσα σήμερα έναν Βρετανό Ευρωβουλευτή που λέει για κάποιες κοινέ διευθετήσεις που υπάρχουν ε, και στην Νορβηγία παραδείγματος χάρη και στην Ελβετία. Θα ήθελα να δω αν υπάρχουν πράγματι διευθετήσεις ε, που βοηθούν αυτές τι χώρε, μάλλον τι ενθαρρύνουν να παραμείνουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση και μήπω και κάποιες χώρε ε, μπουν στον πειρασμό να εγκαταλείψουν την Ένωση για να έχουν τι ε, σχετικέ αυτές διευθετήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις συμφωνίες αυτές υπαρχουν κράτη, κάποια κράτη-μέλη που συνεχίζουν να έχουν πολιτική επιφύλαξη επί της πρότασης και θέλουν να δουν το θέμα ως πακέτο, με προσέγγιση πακέτου, συνδέοντας προτάσεις που τροποποιούν την οδηγία για τις αποταμιεύσεις, για την αμοιβαία συνεργασία, την πρόταση αμοιβαία συνεργασίας δηλαδή, αλλά και την πρόταση που αφορά διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες και κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα θέμα που το επεξεργαζόμεθα και η Βελγική Προεδρία το θεωρεί το θέμα αυτό προτεραιότητα της Προεδρίας της. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσει να σημειώσει πρόοδο σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το θέμα. Τώρα, η... δεν άκουσα την αρχή της δεύτερης ερώτησης. Κύριε Κέλλη, θέλετε να επαναλάβετε πολύ ε, γρήγορα το πρώτο μέρος της ερώτησης, δεν ήταν σαφές. Ένας Βρετανός ε, βουλευτής είπε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση με παρόμοιες ε, δημοσι... Ε, χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις όπως αυτές που έχουν στην Νορβηγία και την ε, Ελβετία. Συμφωνεί η Κομισιόν. Δηλαδή διευκολύνουμε την Ελβετία και την Νορβηγία υπερβολικά, ιδιαίτερα εν ώψη της ερώτησης του κυρίου Παπα-Νικολάου. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση μας απέναντι στις χώρες αυτές, ώστε εκείνες να ενθαρρυνθούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που λένε χώρες καλύτερα να είμαστε έξω από την Ένωση και να είμαστε κι εμείς σαν την Νορβηγία και την Ελβετία. Δεν θέλω να σχολιάσω αν η Βρετανία θα ήταν σε καλύτερη μοίρα μέσα ή έξω από την Ένωση. Αυτό μπορεί κανείς να το δει όπως νομίζει. Αλλά θέματα φοροδιαφυγής, φορολογικών απατών, όλα αυτά τα θέματα. Σε σχέση με την Ορβηγία γίνονται διαπραγματεύσεις με τη χώρα αυτή και έχει γίνει μεγάλη πρόοδο σε αυτό το τομέα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Ορβηγία για αυτά τα θέματα. Και όπως είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία, ζητήσαμε από το Συμβούλιο να μας δώσει διαπραγματευτική εντολή για μια παρόμοια συμφωνία με την Ελβετία. Όμως τώρα είναι τέτοια η κατάσταση ώστε χειριζόμεθα το τωρινό πακέτο που περιλαμβάνει τρεις οδηγίες και το ζήτημα του Λίχτενστάιν και μόνο αφού τελειώσουμε με αυτό το κομμάτι του πακέτου τότε θα μπορέσουμε να πάρουμε εντολή για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με την Ελβετία. και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη όμως δουλεύουμε με την Ελβετία πάνω σε ένα άλλο θέμα, την ε, ισχύ ενός κώδικα δεοντολογίας στη φορολογία των επιχειρήσεων και παρόμοια θέματα και πρόσφατα το Συμβούλιο ζήτησε, μας ζήτησε να αρχίσουμε διάλογο με τις ελβετικές αρχές για να τους βολιδοσκοπήσουμε σχετικά με την εφαρμογή αυτών των αρχών του κώδικα δεοντολογίας στην Ελβετία. Ο, ε, ε, ήδη άρχισε ο Επίτροπος στο διάλογο την περασμένη εβδομάδα και κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορέσω να σας ε, μιλήσω για την πρόοδο που σημειώθηκε. Ευχαριστώ. Η ερώτηση προς την κυρία Τζορτζίεβα. Α, α όχι, όχι, λάθος. Έχει αποσυρθεί η ερώτηση 18 του κυρίου Ζιόμπρο. Και προχωρούμε στην ερώτηση υπαριθμών 19 του κυρίου Πόσελτ. Ο κύριος Φίλε είναι ο επίτροπος που θα απαντήσει. Καλώς ήρθατε, επίτροπε. And ο κανόνας είναι 20 λεπτά ανά επίτροπο, οπότε υποθέτω ότι θα ε, έχουμε τέσσερις από τις ερωτήσεις προς τον κύριο Φίλε μέχρι και την 22. Είμαστε στην ερώτηση 19. Κύριε Φίλε, όταν είστε έτοιμος, μας απαντάτε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει την κατάσταση και τις ανησυχητικές οικονομικές καταστάσεις στη Νότια Σερβία ε, και την περιοχή της κοιλάδας του Πρέσεβο. Ιστορικά η περιοχή ήταν υποανάπτυκτη και ήταν το πιο φτωχό κομμάτι της Σερβίας. Η Κομισιόν έδωσε ε, από το 2000 σημαντική οικονομική βοήθεια στη Νότια Σερβία με στόχο να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ Νότια Σερβίας και της υπόλοιπης χώρας εις ό,τι αφορά συνθήκες διαβίωσης, δημόσιες υπηρεσίες και να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει να ενταχθεί η ε, περιοχή αυτή στους κρατικούς δεσμούς, στο, σχεδιασμό, μελλοντικό, μελλοντικές επενδύσεις ε, και υλοποίησή τους. Για τη διασυνοριακή συνεργασία με το μέσο ΆΙΠΑ για την προενταξιακή υποστήριξη, το πρόγραμμα ε, που αναφέρεται στην ερώτηση θα εξαρτηθεί από την ε, σχέση που θα αναπτυχθεί μεταξύ των εταίρων, των εμπλεκομένων. Εν τω μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει το κράτος δικαίου επενδύσεις, υποδομές και τις ε, τοπικές ε, μεθοριακές ε, συγκοινωνίες μεταφορές. Με τα μέσα που διαθέτει, το τη Γιούλεξ και το, στο Κωσυφοπέδιο και την, το νέο πρόγραμμα, τα νέα προγράμματα ΆΙΠΑ για την Σερβία, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Κωσυφοπέδιο. Τώρα για το Κωσυφοπέδιο τον Οκτώβριο του 2009 οι ανακοινώσεις της Κομισιόν για το Κωσυφοπαίδιο περιλάμβαναν σημαντικές προτάσεις που το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων μας ζήτησε να προχωρήσουμε το Δεκέμβριο. Έτσι το κοσυφοπαίδιο θα αρχίσει ουσιαστικά να ωφελείται από τους πόρους της Ένωσης προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας και αυτό θα γίνει αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους. Θα κινητοποιηθούν συνιστώσα δύο ε, του ΆΙΠΑ για το κοσυφοπαίδιο και την Αλφανία και με τη, γιατί το 2010, φέτος δηλαδή, γιατί ε, το Θα συμπεριλάβουμε το Κωσυφοπαίδιο, το Μαυροβούνιο επίσης του χρόνου. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε αυτό το τομέα μέσα από τον διαρθρωμένο διάλογο με τις αρχές και μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις μας. Η επόμενη θα ε, δημοσιευτεί το Νοέμβριο του 2010. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Πόσελτ, έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την πολύ καλή απάντηση που ε, εσείς είστε από το Regio Εγκρένσης, υποδειγματική περιφέρεια της Ευρώπης και νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, τοπικές μεταφορές ούτως ώστε όταν κάποιος θέλει να πάει στο χωράφι του από την άλλη πλευρά να μην περιμένει μαζί με τους τουρίστες, τουρίστες ε, να μπορεί να υπάρχει αναγνώριση των ε, απολυτηρίων πτυχίων. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και πρέπει να τους δώσετε παρακαλώ προτεραιότητα γιατί ο κόσμος εκεί υποφέρει πολύ. Ευχαριστώ Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, θα είναι προτεραιότητά μου στην περιοχή. Δεν πρόλαβα, δεν είχα χρόνο για να μιλήσω διεξοδικά για τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδιαίτερα στην περιοχή που αναφέρατε. Το θέμα που επισημάνατε ήδη αποτέλεσε θέμα των διαβουλεύσεών μου στο Συμβούλιο Διασυνοριακής Συνεργασίας, το RCC, που αποτέλεσε τη συνέχεια της επιτυχούς συνδιάσκεψης του Σαράγεβο. Ήταν, είναι και θα είναι προτεραιότητά μου λοιπόν στις σχέσεις με τις χώρες αυτές αλλά και τις περιφερειακέ περιφερειακές οργανώσεις που θα μας επικουρήσουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Έχω δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Ο κύριος Τιούντας και ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ο κύριος Χουντή, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ασφαλώς θα γνωρίζετε ότι έχει δημιουργηθεί εκρηκτική κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο από το γεγονός ότι την προηγούμενη Παρασκευή ρίχθηκε χειροβοβίδα εναντίον σέρβων διαδηλωτών που διαδήλωναν κατά της έναρξης λειτουργίας γραφείων της κυβέρνησης του κωσυφοπεδίου στη μητρόβιτσα. επειδή υπάρχει εντός του ιουλίου η απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου της χάγης σε σχέση με την ανεξαρτοποίηση μονομερή ανεξαρτοποίηση του κωσόβου θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή η ενέργεια δηλαδή η ίδρυση γραφείου εξ αντικειμένου έχει προκλητικό χαρακτήρα και θα έπρεπε να είχε αποφευθεί. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Χουντή. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Μισό λεπτό παρακαλώ. Πολύ σημαντικό το ζήτημα της διασυνοριακή συνεργασίας και θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του. Βλέπω όμως και θέλω πραγματικά να το καταγράψουμε αυτό και είναι απαράδεκτο την, ε, ε, την, τον τίτλο στην ερώτηση στον πίνακα, τον επίσημο πίνακα του Κοινοβουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη ονομασία της μιας χώρας από τις τρεις είναι ΦΥΡΟΜ, πρώην ιουγκοσλαβική δημοκρατία της μακεδονίας. Αυτό είναι ο επίσημος ε, τίτλος της χώρας η επίσημη ονομασία και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν και διαπραγματεύσεις μεταξύ ε, της ελλάδας και της ΦΥΡΟΜ για την επίλυση του ζητήματος. δεν είναι δυνατόν σε μια επίσημη συζήτηση να γράφουμε αυτό στον πίνακα του κοινοβουλίου μας. σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα θέλατε να απαντήσετε. Αν μπορείτε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία επιλογής που μου δίνετε να απαντήσω ή όχι. Είχα συνομιλίες με τους δύο πρωθυπουργούς, τον κύριο Κουλαέφηση και τον κύριο Παπανδρέου, και σας διαβεβαιώ μετά από τις συνομιλίες μαζί τους ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για την επίλυση του ζητήματος που επισήμανε ο αξιότιμος Ευρωβουλευτής. Έχουν προχωρήσει αρκετά οι συζητήσεις αυτές και ευελπιστώ ότι οι δύο ηγέτες θα δράξουν την ευκαιρία αυτή προκειμένου να διαθετήσουν το ζήτημα και να, μπορέσουν, να μπορέσει η χώρα αυτή να ξεκινήσει τις ε, ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, πριν από δύο περίπου εβδομάδες βρέθηκα στο βόρειο τμήμα του Κωσυφοπεδίου για τα εγγένεια κοινοτικού γραφείου και μίλησα για το πρόγραμμα και την ανάγκη να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας ε, για τους κατοίκους της περιοχής, για όλους τους κατοίκους, προκειμένου να μην υπάρχουν απομονωμένοι θύλακες. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να αποφεληθούν από αυτά τα προγράμματα. Έχετε απόλυτο δίκιο όμως ε, ότι ε, με βάση την ομολογία του ΔΕΚ θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε πράξη που θα καταστήσει την κατάσταση πιο έκριθμη. Και από αυτή την άποψη, Κάθριν Άστον, είπατε εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά αυτό το τραγικό επεισόδιο, είχε μια τηλεφωνική συνομιλία με ηγέτες ε, και του Βελιγραδίου και της Πρίστινα και πίφθινε έκκληση προς τους ηγέτες των δύο πλευρών να συνεχίσουν την πολιτική εγκράτειας και αποφυγής της βίας. Πολλό δε μάλλον που περιμένουμε να πάσα στιγμή την νομολογία, τη σχετική έκδοση απόφασης. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Θεοχάρου. Ε, δεν είναι παρούσα η κυρία Θεοχάρου, οπότε καταπίπτει η ερώτηση αυτή και περνάμε στην ερώτηση 21 από τον κύριο Χουντή. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να απαντήσετε την ερώτηση 21. Thank you. Uh, Συνεχίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα και σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει την ε, έκκλησή της προς την Τουρκία να εφαρμόσει το πρόσθετο πρωτόκολλο για τη Συμφωνία Σύνδεσης και να άρει όλα τα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ αυτών και περιορισμό των άμεσων ε, εμπορικών σχέσεων με την ε, Κύπρο. Θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει σε σχέση με όλα τα ζητήματα στην επόμενη μάλιστα ετήσια έκθεση θα έχει τα ε, σχετικά στοιχεία, θα προβούμε σε μια καταγραφή των πραγματικών περιστατικών και την πρόοδο ή τη μη πρόοδο στους τομείς αυτούς, όπως κάναμε και πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια. Επί τη βάση αυτή, συγγνώμη κύριε Επίτροπε που σας διακόπτω, αλλά ο κύριος Πόσελτ, επαναλαμβάνω, αν τσακώνεστε, ε, βγάλτε τα ακουστικά σας, γιατί φωνάζετε κύριε Πόσελ, τουλάχιστον βγάλτε τα ακουστικά σας. Διότι διακόπτετε τον Επίτροπο. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να συνεχίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Να επαναλάβω λοιπόν την τελευταία πρότασή μου. Έλεγα λοιπόν ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει με τη βάση αυτή, την έκθεση αυτή λοιπόν να καταλήξει στα κατάλληλα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χουντέ, έχετε το λόγο. Μισό λεπτό παρακαλώ μόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση που μου δώσατε. Θα ήθελα συμπληρωματικά να σας θέσω την εξής ερώτηση. Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστόφιας, συνέδεσε το άνοιγμα των νέων κεφαλαίων της προενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας με το άνοιγμα του λιμανιού της Αμοχώστου, τονίζοντας ότι το λιμάνι μπορεί να παραδοθεί στα Ηνωμένα Έθνη και να λειτουργήσει υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή η ανάλογη πρόταση έχει διατυπωθεί στο παρελθόν το 2006... και είχε θετική ανταπόκριση από τα ηνωμένα έθνη. θα ήθελα λοιπόν να σας πω ποια είναι η γνώμη σας ποια είναι η αντίδρασή σας σε αυτή την πρόταση του κ. χριστόφια. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία είναι επιτάπητος στο πλαίσιο των συνομιλιών για την προσπάθεια εξέβρεσης λύσης ε, στο ζήτημα της Κύπρου. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απολύτως ξεκάθαρος. Όχι μόνο υποστηρίζουμε αυτή την ε, διαδικασία υπό τον ΟΗΕ, όχι μόνο υποστηρίζουμε τους δύο ηγέτες ε, στις προσπάθειές τους για την εξέβρεση λύσης στο Κυπριακό, έχουμε όμως στείλει τον προσωπικό απεσταλμένο του Πρόεδρου της Επιτροπής ε, για να βοηθήσει στην εξέλιξη των συμιλιών μεταξύ των δύο μερών ε, για τα μέτρα αυτά που σχετίζονται όπως είπατε και με τον ΟΗΑ. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα στοιχεία που μπορεί να μην έχουν τεθεί άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά τα οποία είναι σχετικά, διασυνδέονται αν θέλετε με αυτά. Και ένα από τα θέματα αυτά το αναφέρατε μόλις. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι ότι καλεί και τις δύο πλευρές και άλλες χώρες ε, οι οποίες ενδιαφέρονται να είναι δημιουργικές, επικοδομητικές και να καταλήξουν σε μία λύση. Όταν μιλώ λοιπόν για εξέβρεση λύση, συμπεριλαμβάνω και αυτό το ζήτημα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πράγματα. Γιατί αλλιώς το ζήτημα το οποίο εσείς ε, θέσατε ε, θα ενταχθεί ε, στις όλες οι συνομιλίες για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Πριν περάσω στη συμπληρωματική εκ του κυρίου Κέλλη, επαναλαμβάνω, εάν θέλουμε να τελειώσουμε μέχρι τις 8.30 Και το λέω όχι γιατί αυτό προβλέπει η μερίσια διάταξη, αλλά γιατί πρέπει να γίνει και κάποια διακοπή για του διερμηνεί που θα ξαναξεκινήσουν σε νέα. Πρέπει να τηρήσουμε τον χρόνο αγώνα. Ο κύριο Ντεχούχ, το επόμενο επιτρόπο, θα ξεκινήσει γύρω στι 8 και 4. Οι 27, 28, 29. 30 και 31 ε, είναι μη παραδείκτέ. γι' αυτό θα ξεκινήσει ο κύριο Ντεχούχτα με την ερώτηση 32 του κυρίου Ταραμπέλα. Το ερώτημα του κυρίου Κράουλη τώρα. Για τον κύριο Κράουλη δεν έχουμε ενημερωθεί ε, ποιο θα τον αντικαταστήσει. Δεν θα ληφθεί υπόψη λοιπόν και θα περάσουμε στο ερώτημα του κυρίου Χάουιτ. Για μια κοινή απάντηση. Κύριε Γκάλαχερ, θα στείλω κάποιον να σας μιλήσει, ναι. Περνάμε και πάλι λοιπόν στον κύριο Κέλλη, δεύτερη και τελευταία συμπληρωματική. Α, κύριε Μαγκίνες, για διαδικαστικό. Δεν ξέρω αν εσείς θεωρείτε ότι είναι μη παραδεκτά τα ερωτήματα τα δικά μου και άλλων ε, γιατί δεν είναι καλά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι γιατί αφορούν θέματα που είναι στη μέση και της Πέμπτης. Πρέπει να σας πω όμως ότι εμείς δεν γνωρίζαμε ο συντάκτη τη ερώτηση. Εμεί ζητούσαμε να γίνει συζήτηση ε, για τι διμερεί συνομιλίε Μερκοσούρ και γι' αυτό έχουμε Υποβάλλει αυτά τα ερωτήματα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να θεωρηθούν παραδεκτά τα ερωτήματα αυτά. Δεν είμαι μόνη μου, είναι και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν να θέσουν το σχετικό ζήτημα. Θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά απλά για ποιο λόγο έχετε ε, στη συγκεκριμένη ώρα των ερωτήσεων θεωρήσει μη παραδεκτές αυτές τις ερωτήσεις. Κύριε Νίκολς. Δεν σας καθυστερήσω γιατί υπάρχει πίεση χρόνου και το αντιλαμβάνομαι. Συμφωνώ απόλυτα με την προλαλήσασα, την κυρία Μαγκίνες. Και πραγματικά έχω γανακτήσει με τη διαδικασία αυτή. Ξέρω ότι θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε, αλλά το θέμα αυτό είναι φλέγον. Έπρεπε να συζητηθεί και να δοθεί μια απάντηση σήμερα και θα μας βοηθήσει και στη συζήτηση που θα γίνει την, παρασ... την Πέμπτη το πρωί. Φαντάζομαι και οι δύο είστε εμπνευστέ της προφορικής ερώτησης και θα πρέπει να σας συγχαρούμε για τη συμπερίληψη αυτής της προφορικής ερώτησης στο πρόγραμμα της Πέμπτης γιατί έτσι θα έχουμε πολύ ε, καλύτερη ευκαιρία για διεξοδική συζήτηση. Πάντως ευχαριστώ που το επισημάνατε και στο μέλλον θα σας ενημερώνουμε πιο έγκαιρα. Ο κύριος Γκάλαχερ. Το γραφείο μου κύριε Πρόεδρε είχε ήδη ενημερώσει την Προεδρία ότι θα αναπληρώνω εγώ τον κύριο Κρόλη. Ναι, αλλά ο κύριος Κρόλη δεν έκανε την επισήμαση. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Καλά, κύριε Κάλεχερ. Αν έχετε λίγη υπομονή και προλάβουμε, ίσως ε, ασχοληθούμε και με τη δική σας ερώτηση. Κύριε Κέλλη, δεύτερη και τελευταία συμπληρωματική σε ό,τι αφορά την έκθεση Χουντή προς τον Επίτροπο Φίλε. Εμένα με θα με ενδιαφέρει περισσότερο το θέμα των τουρκοκυπρίων αθλητών, γιατί και εγώ αθλητής ήμουν και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν όρια, δεν θα πρέπει να υπάρχουν σύνορα για τους αθλητές. Τα μόνα σύνορα και οι μόνοι περιορισμοί των αθλητών είναι οι δικές τους επιδόσεις. Και έχουμε και το Ολυμπιακό Συμβούλιο. Ε, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε όλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει το Ολυμπιακό Συμβούλιο να επιληθεί. Κρίμα όμω είναι να μπαίνουν περιορισμοί στους αθλητές ο επίτροπο, σα ευχαριστώ. Για το θέμα αυτό, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το θέμα της απομόνωσης των τουρκοκυπρίων αθλητών. Θα πρέπει να επιληθεί μέσω του ενδοκυπριακού διαλόγου και την αναζήτηση μιας ε, γενικότερης λύσης στο Κυπριακό γιατί υπάρχει και το πλαίσιο των Ηνωμένων που προβλέπει τη δυνατότητα αυτών των συνομιλιών, ενώ δεν προβλέπεται αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα πρέπει να επιληθεί το Κυπριακό και ως παρενέργεια θα επιληθεί και το θέμα αυτό των αθλητών. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ηγετών των δύο πλευρών για την ειρηνική επίλυση και ομαλή επίλυση του Κυπριακού κάτι που θα επιλύσει αυτόματα και το πρόβλημα που επισήμανε η Ευρωβουλευτής. Πάντω, οι τουρκοκύπριοι αθλητέ θα πρέπει να αποφασίζουν ελεύθερα σε ποια ομάδα θα, πρέπει να θα μπορούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να υποβάλλονται σε πιέσει ή να υφίσταται πιέσει από οποιοδήποτε πλευρά. Αλλά το θέμα αυτό θα επιληθεί στα πλαίσια του ενδοκυπριακού διαλόγου. Σα ευχαριστώ. Προχωράμε στην ερώτηση 22 του κυρίου Μίτσελ για το Μεσανατολικό. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μείζον παίχτη στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και σε πολιτικό και σε πρακτικό επίπεδο. Σε πρακτικό επίπεδο ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται σε στενές διμερείς σχέσεις με όλους τους εταίρους σε αυτή τη σημαντική περιοχή η πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία αποτέλεσε το πλαίσιο για αυτέ τι διμερείς σχέσεις που μπορεί να προσαρμόζονται προς τις ανάγκες κάθε χώρας. οι συναντήσεις ε, στα πλαίσια της πολιτικής ε, γειτονίας ε, αποτελούν ένα πλαίσιο για πολύ καλές συζητήσεις ε, περιλαμβάνοντας την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποίησε τις συναντήσεις αυτές με το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για να εξετάσει διάφορα θέματα, πολιτικά θέματα, συζητήσεις επί συγκεκριμένων υποθέσεων ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, την κατάσταση επιτόπου, το έργο της υποστήριξής μας και Και κάθε φορά το πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας βοήθησε για να έχουμε τακτή ροή πληροφοριών και ε, ανταλλαγή απόψεων. Σε πρακτικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει σημαντική υποστήριξη για αυτή την περιοχή ως αποτέλεσμα διμερών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει κατά πολύ στις ε, προς προσπάθειες ε, δημιουργίας ε, ε, ενίσχυσης των Παλαιστινίων. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των διμερών σχέσεων με συνέπεια υποστήριξε πολυμερή προσέγγιση για την ειρηνευτική διαδικασία. Η Ένωση για την Μεσόγειο επίσης είναι ένα άλλο πλαίσιο όπου μπορούν να συζητούν όλοι οι εταίροι στην περιοχή. Ε, εις επίμετρον η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείες, τη Ρωσία και τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένα μέλος του κουαρτέτου της τετραμερούς που προωθούν εκ του σύνεγγυ συνομιλίες Ισραηλινών Παλαιστινίων. Στη συνάντηση της 19 Μαρτίου του 2010 η τετραμερής ε, υπέδειξε ότι η Ειρηνευτική Συμφωνία που καλύπτει θέματα καθεστώτος θα πρέπει να συμπληρωθούν μέσα σε, και να ολοκληρωθούν μέσα σε 24 μήνες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίτσελ, ευχαριστώ τον Επίτροπο για την απάντηση. Ε, οι αραβικές χώρες στη Μέση Ανατολή, κύριε Επίτροπε, συνεχώς αποτυγχάνουν να σεβαστούν τις υποσχέσεις τους για την ανθρωπιστική βοήθεια. Μία φορά, νομίζω μέσα της δεκαετίας του 80, δηλαδή μία φορά έγινε αυτό πριν από 20 χρόνια. Οι φορολογούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζορίζονται και ε, θέλουν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις. Γιατί δεν το λέτε. Επίσης έδωσε στοιχεία ο κ. Ντεγκίνγκ, ε, στοιχεία από την Ούνρα, σε μια κοινή συνεδρίαση τριών επιτροπών και είπε ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έκαναν προσπάθειες που κατάφεραν να σκίσουν πιέσεις στην Ισραηλινή κυβέρνηση για την, για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ενώ εμείς δεν το κάναμε. Δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση. Θα είναι δύο κράτη, προσέγγιση δύο κρατών και έχουμε και τον οδικό χάρτη. Ε, δεν πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους στην περιοχή. Ευχαριστώ, ο Επίτροπος. Θα ήθελα, κύριε Ευρωβουλευτά, να ξεκινήσω από εκεί που σταματήσατε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο την ε, ευκαιρία αυτή και να τη διευρύνουμε, γιατί η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή είναι πολύ σημαντική και στο θέμα αυτό συνεργαζόμαστε στενά με την κάθε Άστον, την είπατε εκπρόσωπο και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ευελπιστούμε ότι θα δράξουμε εδώ τους καρπούς ε, της ε, Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής ε, και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όπως διαμορφώνεται μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Με τους νέους μηχανισμούς που έχουμε για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας, είμαι περήφανος που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους σημαντικότερους δωρητές στην περιοχή και είμαι επίσης περήφανος που η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί αυτή την υποστήριξη στη, για την εδραίωση των κρατικών θεσμών του Παλαιστινιακού κράτους. Βέβαια, με προβληματίζει το γεγονός ότι ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα γειτονικέ, δεν ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει και στις, στο επίπεδο συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Μίτσελ, μπορείτε να επαναλάβετε τη δεύτερη σας ερώτηση. Ναι. Θα πρέπει το μήνυμά μας να το μεταδώσουμε με διαφορετικό τρόπο. Ίσως δεν το έχουν καταλάβει μερικές φορές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και μερικές φορές η ειρηνική προσπάθεια επίλυσης ισοδυναμεί με αδράνεια η αναποτελεσματικότητα. Μήπως θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο που μεταδίδουμε το μήνυμά μας. Σας είπα στην αρχή έμεσα βέβαια ότι ναι, όντως χρειαζόμαστε μια καλύτερη επικοινωνία και μια στενότερη συνεργασία με την την εκπρόσωπο και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα πώς θα γίνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο, ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή, στη Μέση Ανατολή. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τους μηχανισμούς της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προκύπτουν μετά τη θέση ισχύ της ηθική Λισαβόνας. Αυτό θα πρέπει να διερευνήσουμε. Ο κύριος Ντέιβις, συμπληρωματική. Ευχαριστώ. Ο ειδικό μα επεσταλμένο Τόνι Μπλερ έδωσε την εντύπωση ότι το Ισραήλ θα άρει, θα χαλαρώσει, θα άρει τον αποκλεισμό τη Γάζα. Από τον Τζον Κίνγκ όμω, τον επιχειρησιακό διευθυντή τη Άντρα, ακούσαμε σήμερα ότι ναι, μεν επιτρέπονται τα τρόφιμα, αλλά δεν μπορεί να το αγοράσει ο κόσμος, ε, διότι δεν μπορεί τίποτε να μπει, δηλαδή είτε για το εμπόριο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο υλοτομέα, ώστε να υπάρχουν έσοδα τον, ε, για τους Παλαιστίνους και να μπορούν να αγοράσουν. Είναι λοιπόν λίγο παραπλανητική και δόλια αυτή η πρακτική. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, τα λόγια και να προχωρήσει σε πράξει. Μέσω τη Συμφωνία Σύνδεση έχει η Επιτροπή τη δυνατότητα να ασκήσει πιέσει στο Ισραήλ. Οπότε θα δούμε λοιπόν πράξει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υπάρξει πραγματικά ανακούφιση στην περιοχή τη Γάζα. Να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ. Επίτροπο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι βέβαιος ότι η Συμφωνία Σύνδεσης ε, και το πλαίσιο αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος ε, να ασκήσει κανείς πίεση σε οποιονδήποτε. Φαντάζομαι γνωρίζετε, αξιότιμα βουλευτά, την προθυμία του Ισραήλ να αναβαθμίσει τις σχέσεις του κράτους Ισραήλ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λεγόμενο advanced status, το προηγμένο αυτό καθεστώς. Λόγω όμως όλων αυτών των ε, αιτίων που ακούσαμε, η αναβάθμιση αυτή δεν έχει ακόμη ισχύσει. Και εμείς βλέπουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάποιες ανεπάρκειες. Αυτό που θέλουμε είναι να λυθεί το ζήτημα του αποκλεισμού της Γάζας. Η Κάθριν Άστον, η Πατή εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος Επιτροπής, καθημερινώς ε, ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Εγώ θα πήγαινα στην ε, περιοχή αυτή. Συμφωνήσαμε όμως με την κάθε Άστον ότι το καλύτερο θα ήταν πρώτα να υπάρξει το άνοιγμα και μετά να μεταβεί στην περιοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δει πώς θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες ε, της περιοχής ε, που είναι πολύ μεγάλες και όχι απλώς ανθρωπιστική βοήθεια. Ο πρόεδρος. Η Βαρόνι Λάτφορντ έχει φύγει και λυπούμε, ε, έπρεπε να της είχα πει, ε, ότι θα μπορούσαμε τελικά να εξετάσουμε και το δικό της ερώτημα. Ο κύριος Ντεχούχτ δεν έχει έρθει ακόμη. θα έρθουμε στο ερώτημα λοιπόν 26 τον ε, συντάκτη του ερωτήματος ε, κύριο Τσαμέσκι ε, τον αντικαθιστά ένας άλλος βουλευτής. Θέλω να ακούσω την απάντηση του Επιτρόπου. Thank you, Mr. Uh... Ευχαριστώ. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και η εφαρμογή των υψηλών προδιαγραφών είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα προσφυλές θέμα. Και μάλιστα έχουμε σχέδια δράσης με τη Γεωργία και το Αζερβαϊτζάν από το 2006 που υπογράφηκαν αυτά τα σχέδια δράση με τις δύο χώρες. Η παρακολούθηση αυτή προβλέπεται στο ετήσιο, στην ετήσια έκθεση προόδου που υποβάλλει κάθε άνοιξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το Αζερβαϊτζάν, η περσινή μας αξιολόγηση κατέληξε σε μία άνηση ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια, σημειώσαμε κάποιες θετικέ εξελίξεις, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε ανησυχίε για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης. Όπως φαίνεται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη 3 η Δεκεμβρίου του 2009. Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία, το 2009 η χώρα σημείωσε σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράση EMP και τι προτεραιότητε, ε, σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου, τι μεταρρυθμίσει ε, του συστήματο απόνομη δικαιοσύνη, τη χρηστή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση τη διαφθορά. Τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, συζητώνται τακτικά στον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε με τη Γεωργία. Ε, συναντήσει έγιναν δύο φορές το 2009 και θα επαραληφθούν οι συζητήσεις αυτή τη βδομάδα στην Τυφλίδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στενές σχέση με τις χώρες αυτές προκειμένου να ε, διαπιστώσει κατά πόσο τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την ΟΑΣΕ. Έχουμε συνεργασία με τις δύο χώρες σε πολλά επίπεδα. Επίσης παρακολουθούμε την πρόοδο που επιτελούν σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις εκθέσεις μας εφαρμογής του σχεδίου δράσης και οι χρηματοοικονομικές πιστώσεις για τις εταιρικές σχέσεις EMP μέσω του μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής Σχέσεις θα αντικατοπτρίζουν από το χρόνο με πολύ διαφανή τρόπο τον τρόπο με τον οποίο τηρούνται οι αρχές του ΕΜΠ e σε θέματα εκδημοκρατισμού, σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Επιπλέον, η ανατολική εταιρική σχέση προβλέπει δυνατότητα νέων και φιλόδοξων ε, συμφωνιών σύνδεσης με τις χώρες αυτές που είναι πρόθυμες αλλά και ικανέ να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις ε, ακόμη και σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βόσεβιτς για συμπληρωματική ερώτηση. Μισό λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ για την απάντηση. Η ερώτηση όμως ήταν αν μπορούν να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα ή κάποιο είδου επιβράβευση στα πλαίσια των δράσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενθαρρυνθούν αυτοί που πληρούν τα κριτήρια και τις προδιαγραφές και να επιβραβευθούν με συγκεκριμένες αντισταθμίσεις. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα παροχής κινήτρων σε αυτούς που τηρούν τις προδιαγραφές. Ο κύριος Επίτροπος. Συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή ότι η πολιτική γειτονίας προωθεί τις μεταρρυθμίσεις. Οπότε όσο πιο προσιλωμένες οι μεταρρυθμίσεις η ε, εταίροι μας, τόσο πιο δραστήρια και ενεργά θα πρέπει να υποστηρίξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χώρα αυτή στις προσπάθειες ε, τις μεταρρυθμιστικές. Και αν ρίξετε μια ματιά στις ε, χώρες που συμμετέχουν στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, διαπιστώνεται ότι Όντως είναι αποτελεσματική αυτή η πολιτική. Και αποφέρει καρπούς. Έχουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης, τη Συμφωνία Οικονομικής Ολοκλήρωσης και το θέμα της ε, κινητικότητας ε, ή των θεωρήσεων ή συναφή ζητήματα. Αν δείτε λοιπόν πόσες χώρες συμμετέχουν στην ανατολική εταιρική σχέση, βλέπετε πόσο διαφορετική είναι η στάση τους απέναντι στις μεταρρυθμίσεις και πόσο διαφορετική είναι και η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στις χώρες αυτές. Και η Μολδαβία είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με τη χώρα αυτή ξεκινήσαμε αρχικά τις διαπραγματεύσεις ε, για συμφωνία προσχώρησης και με τη χώρα αυτή αρχίσαμε και το διάλογο για τις θεωρήσεις. Και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα οι χώρες αυτές θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και οικονομικής ε, ολοκλήρωσης και ελεύθερο εμπορίου. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα στις ερωτήσεις προς τον κύριο Ντεχούχτ. Ήρθε στο μεταξύ κυρία Μαγκάβαν και χαίρομαι ιδιαίτερως. Ο κύριος Ταραμπέλα δεν είναι στη θέση του, οπότε καταπίπτει η ερώτησή του. Αλλά προβλέπεται κοινή απάντηση στις ερωτήσεις ε, Ταραμπέλα και Μακάβαν. Ο κύριος Ντεουκχούχτ έχει το λόγο. Για τις ερωτήσεις 32 και 33. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το δίκαιο εμπόριο και όλα αυτά τα συστήματα έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την προώθηση ε, της εξέλιξης και για τις ενημερωμένες επιλογές καταναλωτών. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι είναι μη κυβερνητική Όπω χαρακτήρα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Μαΐου 2001 για αυτά τα συστήματα, θα πρέπει η κυβερνητική παρέμβαση να είναι περιορισμένη ώστε να μην αναμειγνύονται στο δυναμικό χαρακτήρα του δίκαιου εμπορίου και των προτιμήσεων των καταναλωτών. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχει πρόβλημα, ενδέχεται να υπάρξει σύγχυση ε, των καταναλωτών, γι' αυτό Διάφοροι φορείς όπως ε, το Διεθνώς Εμπορικτό Κέντρο η UNCTAD ε, θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούν να βοηθήσουν ε, καθιστώντας πιο διαφανή και σαφή τα κριτήρια. Σε ό,τι αφορά την ευθύνη τη Επιτροπή για συστήματα δίκαιου εμπορίου, η Επιτροπή έχει, ευθύ... έχει χωρίσει την ευθύνη σε διάφορου επιτρόπου. Παραδείγματο χάρη, τα Γιάννη και Μπαρνιέ είναι αρμόδιοι για την εκπόνηση του οδηγού για κοινωνικά υπεύθυνους διαγωνισμούς, ε, τάλι για την ενημερωμένη πλήρη καταναλωτών και πίμπαλξ για σχέδια σε αναπτυσσόμενε χώρε. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπόριο διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό συντονιστικό ρόλο επί του παρόντο, ώστε οι πρωτοβουλίε, οι πολιτικέ να είναι συνεπεί, συνεκτικές με την ανακοίνωση του 2009. Και θα ήθελα να πω ότι θα συνεχίσω ε, ε, το έργο του προκατόχου μου σε ό,τι αφορά αυτόν τον συντονισμό και το ρόλο της Επιτροπής. Η κυρία Μάκαβαν για συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ακούω ότι θα συντονίσετε. Οπότε θα υπάρχει ε, μια σύνδεση των υπηρεσιών σας με τα θέματα του ε, δίκαιο εμπορίου. Χρειάζεται συντονισμό και με τον Επίτροπο Βαρδιέ, γιατί πριν από λίγε εβδομάδε υπήρχαν διατυπώσει στο κείμενο που θα είχε βλάψει το ε, δίκαιο εμπόριο. Ευτυχώ ο Επίτροπο Μπαρνιά παρενέβη, αλλά υπάρχει μια έλλειψη συνοχή με το παλιό κείμενο. Ε, θα είναι συντονιστική ομάδα δηλαδή, η υπηρεσία σα. Συνδέστε με όλε τι διάφορε υπηρεσίε και πώ αυτό λειτουργεί στην πράξη. Ευχαριστώ. Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε, αυτό θα γίνει βέβαια σε επίπεδο διυπηρεσιακό και θα φροντίσουμε να γίνεται συντονισμός με τους άλλους επιτρόπους σε τακτά διαστήματα και έτσι μέσα από αυτό το συντονισμό θα ε, βγει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα και αν χρειαστεί θα κάνω και απευθεία συνομιλίες με τους συναδέλφους ε, επιτρόπους. Ευχαριστώ για τη συντομία σας ε, κύριε Επίτροπε. Πάμε... Α, καταπίπτει 34 ερώτηση, αλλά ο επόμενος παρόν Ευρωβουλευτής είναι ο κύριος Χάουιτ. να είστε σύντομοι παρακαλώ πολύ, γιατί Είπα ότι πρέπει να τελειώσουμε στις 8.30 αφού οι διερμηνείς πρέπει να φάνε κάτι πριν επανέλθουν στις 9. Ε, ε, ερώτηση λοιπόν 35-36 των κυρίων Χάουιτ και Μάρτιν. Έχετε το λόγο. Πολύ σύντομα πράγματι κύριε Πρόεδρε γιατί αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε διαμακρό να συζητήσουμε να πω μόνο ότι οι διαπραγματεύσει σε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με Κολομβία και Περού ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, αλλά η συμφωνία ακόμη δεν έχει μονογραφηθεί επισήμω. Το κείμενο τώρα εξετάζεται από νομικού για να υπάρχει συνοχή ε, και συνέπεια των κειμένων στα αγγλικά και στα ισπανικά. Το φθινόπωρο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και αφού οι διαπραγματευτές το μονογραφήσουν θα υποβληθεί για να υπογραφεί από το Συμβούλιο και το FTA θα ε, υποβληθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σύμφωνη γνώμη μετά την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή. Σε αυτό το στάδιο είναι δύσκολο να προβλέψουμε πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. Μάλλον όμως θα γίνει το δεύτερο εξάμεινο του 2011 δεν είναι σαφέ αν τα εθνικά κοινοβούλια θα κληθούν επίση να εγκρίνουν τι συμφωνίε Η Κομισιόν θα εξετάσει αν χρειάζεται επικύρωση από τα κράτη-μέλη όταν ε, πάρει την οριστική μορφή το κείμενο, λαμβάνοντα υπόψη τη νέα κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Μπορώ να πω ότι υπάρχει και μεγάλη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή αυτό είναι ουσιώδες σημείο των σχέσεών μας, μπορεί να οδηγήσει λοιπόν σε περίπτωση παραβίωσης στην ε, ε, μονοπλευρή διακοπή της συμφωνίας. Αυτό θα γίνει με απόφαση που θα ληφθεί με ειδική πλειοψηφία από το Συμβούλιο με βάση πρόταση είτε της Κομισιόν ή της ΥΠΑ της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της ΚΕΠΑ με βάση το 218.9 της Συμφωνίας της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης. Το κείμενο μαζί με τα ανθρώπινα δικαιώματα θα υποβληθεί στην Επιτροπή ΙΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Χάουιτ και μετά ο κύριος ε, Μάρτιν. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Επιτρόπε, για την απάντηση. Γνωρίζετε τα τελευταία ε, έγγραφα ε, από την υπηρεσία πληροφοριών από την Κολομπία που δείχνουν ότι υπήρχαν παράνομες δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών στην Ευρώπη κατά μιας βελγικής οργάνωσης ε, και της Amnesty International. Δηλαδή αυτές είναι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό συζητήθηκε στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι σημαντικές και σοβαρέ πληροφορίε αυτές που πρέπει να διερευνηθούν γιατί αυτό είναι σημαντικό για το τι θα κάνουμε ε, από εδώ και πέρα ε, με το σχέδιο Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών με την Κολομβία. Ευχαριστώ. κύριος Μάρτιν. Είπα εκπρόσωπος είπε ότι είναι σημαντικό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι αξιολόγηση έχει γίνει, κύριε Επίτροπε, της πιθανής αντίδρασης της Κολομβίας από την Συμφωνία FDA. Ε, θα βοηθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ενδεχομένως θα τα βλάψει. Αναφέρθηκε ότι υπάρχει μια ρήτρα αναστολή. Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά πριν υπογράψουμε θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα προωθηθούν με αυτή τη συμφωνία τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα ε, πάνε πίσω. Έχει γίνει μια τέτοια αξιολόγηση ο Επίτροπος. Ευχαριστώ. Καταρχάς, για την υποτιθέμενη κατασκοπία των μυστικών υπηρεσιών της Κολομβίας. Γνωρίζουμε τις ε, φήμες αυτές και θα τις διερευνήσουμε. Και μάλιστα στο διάλογο με την Κολομβιανή Κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε αυτό το θέμα και στην πρόσφατη ε, επίσκεψη του Μαρτίου του 2010 του Γενικού Διευθυντή αλλά και στις επαφές που έχουμε στο γραφείο μας στην Πογκοτά με το Αρμόδιο Υπουργείο και άλλα υπουργεία τη Κολομβιανή κυβέρνηση και θα παρακολουθήσουμε το ζήτημα εκ του σύνεγγυ για να δούμε αν όντω υπάρχει τέτοια είδου κατασκοπία από τι μυστικέ υπηρεσίε τη Κολομβία σε ευρωπαϊκό έδαφο. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κ. Μάρτιν, όντω έγινε αυτή η αξιολόγηση και σε τελική ανάλυση η αξιολόγηση είναι πολιτικού χαρακτήρα. Γνωρίζουμε ποια είναι τα μέσα που έχουμε και είναι τα σωστά, αλλά πριν μιλήσουμε για μέσα και προσφυγές ή διορθώσεις, θα πρέπει να να δούμε αν όντω η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου θα ενισχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή θα τα παρεμποδίσει. Η δική μου πολιτική αξιολόγηση είναι ότι δεδομένη τη γενική κατάσταση της Κολομβίας η σύναψη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου θα αποβεί προ όφελο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε και ευχαριστώ συνάδελφοι για τι ερωτήσει σα. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίο βέβαια ε, κανονικά είναι απόλυτα αμερόληπτος και αντικειμενικός, αλλά ελπίζω να κερδίσει η Ολλανδία σήμερα στον αγώνα. Διακοπή τη Συνόδου μέχρι τις 9.